πώς θα κερδίσουμε την πρόκληση για το μέλλον και πώς θα οικοδομήσουμε μια δυνατή Ισπανία σε μια ένωση πρωταγωνιστή. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. Ολοκληρώνουμε δηλαδή την ημερήσια διάταξη για τη σημερινή συνεδρίαση. Αύριο, 5η, 3 Φεβρουαρίου 2011, έχουμε συνεδρίαση από τι 9 μέχρι, τις, μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Τα πρακτικά είναι στη διαθέση σα στο ε, δικτυακό χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου